Ε, δέχεστε την ημερήσια διάταξη για αυτή την ε, συνεδρίαση, αντιρρήσει, όχι, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι η συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν το ΕΦΣΥ εγκρίθηκε από την διάσκεψη των Προέδρων και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στη συνέχεια θα, μετα... θα διαβιβαστεί στα μέλη. Έχω δε το προνόμιο να ε, καλωσορίσω σήμερα μεταξύ μας τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν, τον οποίο χαιρετίζω και εξ σας και στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο. Σας θυμίζω επίσης ότι δύο συνεισηγητές ε, αποφάσισαν να επιταχύνουν το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες μας αυτές όσον αφορά το FC2 που είναι σαφής ε, προτεραιότητα πολιτική για όλα τα, τους θεσμούς έτσι ώστε το φάκελος αυτός να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί πριν το πέρας της Μαλτέζικης Προεδρίας. Γι' αυτό και θα δώσω αμέσως το λόγο ε, στον Αντιπρόεδρο Κατάινεν για την εισήγησή του που θα διαρκέσει γύρω στα 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον, ε, στους εισηγητές για 5 λεπτά ο καθένας και στη συνέχεια θα δώσω την, τον λόγο στους κοιόδης ε, για εναλλάσσοντας τους τη ε, της ΕΚΟΝ και της Budget. Θα δώσω λοιπόν ε, τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Επίσης, ε, έχω σκοπό να μιλήσω για το ε, εύση όπως είναι και την πιθανή του παράταση. Και ενδιαμέσως θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα που θεωρώ πως είναι κέρια. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του υφιστάμενου εύση. Εξακολουθεί να είναι η έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης. Δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει καν ε, για το ΕΦΣΙ και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Έχουμε δει και συμμετάσχει σε εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο στις περιφέρειες διαφόρων χωρών που εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από ευρωβουλευτές και που αφορούσαν το ΕΦΣΙ. Ε, αυτές, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις είναι εξαιρετικά καλές και σας ενθαρρύνω να οργανώνετε τέτοιες εκδηλώσεις μαζί με τους συνεργάτες μας της Κομισιόν αλλά και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις πρωτεύουσές σας αλλά και στις περιφέρειες γιατί ε, Πρέπει να συνεχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους επιχειρηματίες, τις τράπεζες, τις τοπικέ αρχές και να εξηγούμε διαρκώ τι είναι το ΕΦΣΙ καθώς και να του δίνουμε καλά παραδείγματα για το τι έχει ήδη πετύχει το ΕΦΣΙ ή πώς έχουν ε, χρησιμοποιήσει το ΕΦΣΙ άλλε περιφέρειε, περιφέρειες, σε άλλες αρχές ή άλλοι ιδιώτε. Διαφορετικά, ε, κατά τα άλλα, το ΕΦΣΥ τα πάει πάρα πολύ καλά και θα σα δώσω και τα τελευταία στοιχεία για το ΕΦΣΙ. 197 προγράμματα υποδομών έχουν πάρει χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ. Αυτά τα projects αντιπροσωπεύουν έναν όγκο χρηματοδότησης 24 δις, πάνω από 24 δις. 24 δις λοιπόν από το ΕΦΣΥ έχουν πάει στην χρηματοδότηση 197 προγραμμάτων ε, ε, υποδομών και καινοτομία. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει εγκρίνει 264 μικρές και μεσές συμφωνίες χρηματοδότησης με τοπικές ε, ή μικρές τράπεζες με χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 8 δις ευρώ. Ως αποτέλεσμα, περίπου 400.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν. 400.000. Πάρα πολλές. Αυτό το παράθυρο λοιπόν για τις μικρομεσαίες θα πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης, αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε ήδη

που από κοινού συγκεντρώνουν μικρές και μεγάλες επενδύσεις. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο και μικρότερα project ε, υποδομών ή καινοτομίας μπορούν να ωφεληθούν από το ΕΦΣΥ. Βεβαίως χρειάζεται όπως είπαμε, να ε, υπάρξει περισσότερη ενημέρωση και να βοηθηθούν τα κρατημέλη, τοπικές αρχές, αλλά ακόμα και ο ιδιωτικό τομέα να δημιουργηθούν έτσι περισσότερες πλατφόρμες, γιατί είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να χορηγηθούν πόροι και σε μικρότερα έργα. Ε, επίσης, υπάρχουν κάποια παραδείγματα από projects όπου η χρηματοδότηση έχει προέλθει όχι μόνο από το ΕΦΣΥ αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα υπόρους της Ένωσης όπως από τα Διεθνωτικά Ταμεία ή από το Horizon ή από το Συνδέοντα στην Ευρώπη. Και αυτά, αυτό είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας για φέτος, για την Κορίνα Κρέτσου και μένα, που θέλουμε να βοηθήσουμε κυρίως τις τοπικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές να συνδυάσουν το ΕΦΣΙ με άλλα ταμεία ευρωπαϊκά, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να μοχλεύσουν ε, και διαρθωτικά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανομή, το ΕΦΣΙ καλά τα πάει επίσης. Αν κοιτάξουμε τις χώρες οι οποίες έχουν υποφεληθεί περισσότερο από το ΕΦΣΥ, οι, μεγαλύτερες, οι μεγαλύτεροι αποδέκτες είναι η Εστονία, Βουλγαρία 2, Ισπανία τρίτη χώρα, Λιθουανία και Πορτογαλία πέμπτη. Η Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, είναι η έκτη. Αν δείτε τι επίπτωση είχε η χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ ανά ΑΕΠ, αυτή είναι. Πολλοί βλέπουν τα νούμερα ως εξή. Πόσα προγράμματα, πόσα project έχει κάθε χώρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πόσα project εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το ΕΦΣΙ αναχώρα. Δίνει κάποιες απαντήσεις και αυτή η κατανομή, αλλά δεν μιλάει για την επίπτωση του ΕΦΣΙ στο ΑΕΠ. Αν θες να μετρήσεις πόσο αποτελεσματικό ήταν το ΕΦΣΙ σε διάφορες χώρες θα πρέπει να κοιτάξει την επίπτωσή του στο ΑΕΠ ή στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και υπάρχει την έννοια τα πάει καλά το ΕΦΣΥ. Πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αλλά ακόμα και τώρα δεν έχουμε σωστή, απόλυτα σωστή γεωγραφική κατανομή. Υπάρχουν διάφορες χώρες ε, ακόμα που για διάφορους λόγους δεν έχουν χρησιμοποιήσει το ΕΦΣΥ παρότι υπάρχει ζήτηση για τέτοια χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να κατηγορήσω κανένα, αλλά για να συγκρίνουμε δύο χώρες ε, που είναι γειτονικέ, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Βουλγαρία, όπως σας είπα, είναι η δεύτερη χώρα που υποφελήθηκε από το ΕΦΣΥ. Βλέποντα την επίπτωσή του στο βουλγαρικό ε, ΑΕΠ ενώ η Ρουμανία είναι η πρώτη τελευταία. Και χρησιμοποίησα πολύ λίγο το έψι. Ποιο είναι ο λόγο για αυτή τη διαφορά. Ένα λόγο είναι ότι στην Βουλγαρία οι τράπεζε ήταν πολύ ενεργέ ε, και χρησιμοποίησαν το έψι. Υπάρχουν ε, τρει ή τέσσερι συμφωνίε μεταξύ των ε, τραπεζών που εδρεύουν στη Βουλγαρία και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που στηρίζεται από το ΕΦΣΥ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης διάφορα ε, έργα υποδομών που έχουν υποφεληθεί εκεί από το ΕΦΣΥ. Ενώ στη Ρουμανία όταν πήγα τελευταία φορά μίλησα με τις μεγαλύτερες τράπεζες ε, της Ρουμανίας ε, και μίλησα για αυτή την υποχρησιμοποίηση και τους λέω γιατί δεν χρησιμοποιεί το ΕΦΣΥ. και μου είπαν ότι δεν υπάρχει ζήτηση για χρηματοδότηση στη Ρουμανία. Τους είπα ότι αμφιβάλλω. Αλλά προφανώ εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, τους λέω. Ενδιαφέρον πάντως, γιατί οπουδήποτε αλλού η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, απαιτεί μεγαλύτερη υποστήριξη. Αυτή ήταν μία από τι εξηγήσει. Οι τράπεζε στη Ρουμανία δεν προσέφηκαν στο ΕΦΣΥ. Δεν χρησιμοποίησαν το ΕΦΣΥ. Ένα άλλο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησε το ΕΦΣΥ, η προηγούμενη ρουμάνικη κυβέρνηση δεν ε, κληρονόμησε, ας πούμε, τιμοπαράδοτα σχέδια, έτοιμα δηλαδή προς χρηματοδότηση. Δεν ήταν όριμα αρκετά τα project. Γι' αυτό οι δημόσιες αρχές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μαζί με τον ιδιωτικό τομέα το ΕΦΣΙ για να χρηματοδοτήσουν ε, project ε, υποδομών. Αλλά αυτό δεν προδικάζει και το μέλλον. Εμείς χρησιμοποιούμε το... τα κρατη να χρησιμοποιήσουν το ΕΦΣΙ ε, στις χώρες συνοχής ε, και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο προσπαθούμε να, να βοηθήσουμε τις χώρες και τις τοπικές αρχές για να χρησιμοποιήσουν το, το ΕΦΣΥ. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε και τη γεωγραφική κάλυψη και θα πάει το ΕΦΣΥ και τα λεφτά του ΕΦΣΥ σε χώρες που οι χρηματακόρες δεν είναι πολύ καλά, πολύ προετοιμασμένες, πολύ όριμες κτλ. Δύο λόγια ε, για το μελλοντικό ΕΦΣΥ 2.0. ξέρετε διάφορα πράγματα γι' αυτό, δεν θα τα ξαναπώ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την προσθετικότητα. Και η προσθετικότητα θα πρέπει να βελτιωθεί σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Καλή είναι και σήμερα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τη βελτίωσή της. Ένας τρόπος για να τη βελτιώσουμε είναι να αυξήσουμε τη διαφάνεια των αποφάσεων. Θα σταματήσω εδώ και είμαι σίγουρος ότι χάρη σε ερωτήσεις σας θα πάρει αυτή η συζήτηση την τροπή που θέλετε. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσίασή σας. Πολύ αισιόδοξη από τη μία, από την άλλη όμως υπογραμμίζει και τις αδυναμίες του ΕΦΣΥ και τα σημεία που πρέπει να βελτιωθεί. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο συνεισηγητές τον κύριο Φερνάντε και στον κύριο Μπούλμαν, ο καθένας για πέντε λεπτά. Όποιο θέλει, ξεκινάει πρώτος. Ο κύριος Φερνάντε. Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ε, σας ευχαριστώ που μου είπατε κύριο ε, Πρόεδρο. Θέλω να χαιρετήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής και όλους τους συναδέλφους. Όντως το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων λειτουργεί καλά, αλλά θα μπορούσε να ε, ε, λειτουργήσει καλύτερα. Και από εκεί προκύπτει όλη η συζήτηση και όλες οι προτάσεις που έχει υποβάλει η κάθε πλευρά. Ε, θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να περάσουμε τα 500 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια καλή γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων αυτών, να είναι προσθετικό, αλλά και, να είναι συμπληρωματικό, αλλά να είναι και καθολικό για όλους. Ε, και ξεκινώ από την παραπληρωματικότητα. Συμπληρωματικότητα δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά συμπληρωματικότητα στις διαφορετικές περιοχές, ούτε όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του project του κάθε project ούτε και όσον αφορά ε, την απόδοση. Δηλαδή, ένα project 50 εκατομμυρίων ευρώ στο Βερολίνο δεν θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο όπως στη Λισαβόνα, αλλά 50 δισεκατομμύρια στη Λισαβόνα δεν ε, θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο όπως σε μια πιο φτωχή περιφέρεια. Η συμπληρωματικότητα λοιπόν δεν μπορεί να είναι αντίθετη ε, να, έχει, ε, να περιμένουμε να έχει τον ίδιο αντίκτυπο όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη, αλλά να βλέπουμε κάθε φορά την ίδια την περιοχή, την ίδια την περιφέρεια, ε, ανάλογα αν είναι πλούσια ή φτωχή. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι ο κίνδυνο μάλλον για ένα ίδιο σχέδιο, για ένα ίδιο έργο δεν είναι ο ίδιο σε όλα τα κατημέλη και ούτε ο ίδιο σε όλα τα ε, τις περιφέρειες ακόμα και στο ίδιο κράτος. Γι' αυτό και θα έπρεπε από ε, την κάθε πλατφόρμα να περιμένουμε διαφορετική απόδοση. Και είναι σημαντικό για να προσθέσουμε, να, να, να αυξηθεί η ζήτηση, να αυξηθεί η ποιότητα των project, ε, να βοηθήσουμε Ακόμα και αν υπάρχουν ήδη 21 πλατφόρμες, πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερες πλατφόρμες, ε, τόσο όσον αφορά αυτές που καλύπτουν τα project ή πλατφόρμες που μπορούν να δουλέψουν, ας πούμε, στον τομέα της ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία για να μπορέσει να κινηθεί σε διάφορα κράτη-μέλη στον τομέα της ενέργειας, ας πούμε. Ένα παράδειγμα δίνω. Θα μπορούσαν να Απέξουν λοιπόν τα κράτη-μέλη μια ε, δραστήρια, μια ενεργητική στάση, ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε συνέργειες ανάμεσα στις τοπικές και τις εθνικές αρχές και είναι σημαντικό και οι τράπεζες που ε, προωθούν και αλθώς και οι θεσμοί χρηματοδοτικοί ή αναπτυξιακοί να είναι ενεργό μέρος όλης αυτής της προσπάθειας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερη γεωγραφική κάλυψη, με μικρότερα project, έτσι ώστε, μάλλον, τότε ενδιαφέρον για να επιτευχθεί αυτό ένα κομμάτι των εγγυήσεων να ε, γίνεται, δίνεται μέσω αυτών, αυτής της πλατφόρμας κάθε φορά ώστε να μπορέσουμε πλήρως να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό αυτού του ΕΦΣΥ. Τώρα, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μικρά, διάφορα πολλά μικρά προγράμματα που μαζί μπορεί να φτάσουν σε ένα σημαντικό ποσό. Ε, γι' αυτό η πλατφόρμα θα μπορούσε να παίξει τον πυρήνα εντό του οποίου να τοποθετηθούν και αυτά τα μικρά τράπεζα. Και γι' αυτό είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Και γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο αυτέ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν μεγαλύτερη, καλύτερη θέση όσον αφορά το παράθυρο των επενδύσεων. Ενώ οι μικρές μικρές επενδύσεις δεν διοχετεύονται μέσω του παράθυρου των επενδύσεων, αλλά μέσω του παράθυρου των μικρομεσαίων, ε, ενώ περιμένουμε και την παρέμβαση των εθνικών και εμπορικών τραπεζών. Βεβαίω και σε αυτό συμφωνούμε, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια τόσο όσον αφορά την Επιτροπή των Επενδύσεων όσο και τον τρόπο επιλογής ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει μια στάση λογική. Τώρα, όσον αφορά τους ηγητές, εγώ είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον συνάδελφο ε, Μπούμερ, ότι δηλαδή θέλουμε να επιταχύνουμε συμφωνούμε ότι θέλουμε να, να, να επιταχύνουμε αυτή την παράταση της νομοθεσίας και μάλιστα όπως είπα να ολοκληρωθεί η συσχετική συζήτηση εντός της Μαλτέζικης Προεδρίας δηλαδή τον ε, Ιούνιο. Και τήρησα το χρόνο μου. Πρόεδρε, πέντε λεφτά, τέλεια. Ε, θα δώσουμε το λόγο τώρα στο συνάδελφο Μπούλμαν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και να σας πω το εξής. Οι δύο συνεισηγητές, ο φίλος μου Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, μας ε, μοίρασαν την έκθεση. Και έτσι λοιπόν, μοίρασαμε την ε, έκθεση αξιολόγηση και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με του ε, εισηγητές και του κοιόδους εισηγητές και όλε τι πληροφορίε από την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ο αντιπρόεδρο λοιπόν ε, Κατάινεν βρίσκεται εδώ και τον ευχαριστούμε που συμμετέχει σε αυτή την άσκηση. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ απευθύνομαι προ τα άλλα θεσμικά όργανα. Την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε με του συναδέλφου, βλέπετε. Και θα ήθελα να πω λοιπόν το εξή. Πιστεύω, και αυτό φάνηκε και στο FC1 άλλωστε ήδη, ότι δεν υπάρχει κανένας τόπος στην Ευρώπη όπου το σχέδιο αυτό το επενδυτικό ακολουθείται με τόσο μεγάλη δέσμευση όσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαστήκατε έξι μήνες για να καταρτήσετε το σχέδιο για το ΕΦΣΥ. Εμεί στη συνέχεια σε λίγες εβδομάδε καταφέραμε να προχωρήσουμε τα πράγματα για το νομοθετικό αυτό σχέδιο. Και κύριε Αντιπρόεδρε, είναι ένα θέμα κριτική αυτό σε ό,τι αφορά την νομοθεσία μεταξύ Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, όπου εσεί ε, κατά 80% βρίσκεται συνένεση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Ήταν λοιπόν πραγματικά ασυνήθιστο αυτό και είμαστε διατεθειμένοι να δείξουμε εκ νέου τέτοια προθυμία και δέσμευση με απόλυτη πεποίθηση γιατί θέλουμε να ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες και ξέρουμε ότι οι δικές και αναλύσεις καταδεικνύουν ότι σε κάποιους τομείς έχουμε έλλειμμα επενδυτικό 200 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη ανά ετός. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να επιτρέψει το FC1 ούτε το fc να είναι ανεπαρκή. Γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε δίκαιο σε όσους επικρίνουν και όσους ε, εξαγάγουν το συμπέρασμα ότι δεν ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα. Δεν θα επιτρέψουμε οι γραφειοκρατικές λεπτομέρειες ε, λοιπόν μοντέλων ή λόγω έλλειψης συνεργασίας, αν θέλετε, και έλλειψης θέλησης συνεργασίας να οδηγήσουν σε αποτυχία το ΕΦΣΥ. Πού βρίσκονται λοιπόν τα προβλήματα και αυτό το παρουσιάσαμε εκτενώς στην έκθεση αξιολόγησης. Έχουν σημειωθεί πολλές επιτυχίες, μεν, σε ό,τι αφορά την ποσοτική παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά υπάρχουν και ερωτηματικά. Και εσείς το είπατε. Μιλήσατε για την συμπληρωματικότητα, για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το ΕΦΣΙ να κατηγορηθεί ότι ένα τμήμα των επενδύσεων προκαλείται από ουσιαστικά αντικατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών επενδύσεων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε και το ΕΦΣΙ και η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα να συνεργάζονται επαρκώς σε ό,τι αφορά το μοντέλο των τιμών και τη μορφή της συνεργασίας. Το ανέφερε ο συνάδελφος Φερνάντες ότι τα πιο σημαντικά και ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα μικρομεσαία εγχειρήματα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν στην διάρθρωση του ΕΦΣΥ να εξετάζουν μόνο ε, project 50 εκατομμύρια και άνω. Για τον απλό λόγο ότι η Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί ότι θα πρέπει να τα επενδύει όλα, να τα ελέγχει όλα και δεν ε, ε, εμπιστεύεται ούτε τις πλατφόρμες, ε, ούτε και τις τοπικές, ε, τα τοπικά θεσμικά όργανα και τις τοπικές τράπεζες. Μίλησατε για 21, για πλατφόρμες. Είναι ένα καινούριο Α, συμπέρασμα αυτό. Και θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά, γιατί τελικά θέλουμε να διοχετεύσουμε τα χρήματα στα εγχειρήματα εκείνα, στα project εκείνα, όπου κρύβεται το μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό το είπε και ο κύριος Πρόεδρος, το είπε και ο συνεισηγητής μας, ο συνεισηγητής μου. Θα εργαστούμε γρήγορα, αλλά ένα σήμα προς το Συμβούλιο. Δεν φτάνει μόνο να συνενέσει γρήγορα. Θα πρέπει να κατανοήσει και γρήγορα το ζήτημα και να προσπαθήσουμε από κοινού να επιλύσουμε τα προβλήματα. Μόνο τότε θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο που θα ήταν να ολοκληρώσουμε όλα αυτά μέσα στην Μαλταϊσική Προεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω το λόγο στον σκιώδη, στους σκιώδης για δύο λεπτά, ευκρινίζω, δύο λεπτά. Και δυστυχώς, ε, το λέω και σας προειδοποιώ, θα είμαι αυστηρός. Ο κύριος Ότμαρ Κάρας, λοιπόν. Α, συγγνώμη. Όχι, όπως τα λέτε η συνάδελφος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ τα δύο λεπτά. Οι δύο εισηγητέ ούτω ή άλλω μίλησαν για όλε τι ανησυχίε και αμφιβολίες που έχουμε σε αυτέ τι δύο επιτροπέ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ενημέρωση. Ο αντιπρόεδρο Κατάινεν το είπε ότι Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι το ΕΦΣΙ. Πολλοί μιλάνε για το σχέδιο Juncker, αλλά δεν ξέρουν αν είναι επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε πολύ πιο κοντά στους πολίτες. Η Κομισιόν έκανε πολλές προσπάθειες, το ξέρω, για να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται στην πραγματικότητα ε, για αυτό το ΕΦΣΙ. Για το θέμα της ε, προσθετικότητας, το έχουμε πει χίλιες φορές, θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά αν θέλουμε να αυτό συνδέεται με την ε, διαφάνεια. Γιατί πολλέ φορέ οι αμφιβολίε που υπάρχουν για την θετικότητα είναι δεν ξέρουμε τι αξία έχει, πώς αξιολογήθηκε το project και πόσο συμμετέχει το ΕΦΣΙ, πόσο συμμετέχει δηλαδή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Μερικές φορές ε, θεωρούμε ότι το τάδε project, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά όταν έχουμε τα στοιχεία, μερικές φορές μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη. Επομένως, πρέπει να φτιάξουμε αυτές τις πλατφόρμες και επίσης ε, είναι σημαντικές αυτές οι πλατφόρμες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Ε, έγινε η πρόταση για μείωση κατά 35% ε, του ποσού της εγγύηση. Ε, δεν ξέρω. Προφανώς η Κομισιόν θα σε εκπλήξει ότι δεν είναι, χαιρόμαστε που πάει χρήμα από το Connecting Europe Facility για να, χρηματο... για να τροφοδοτήσει, αν θέλετε, αυτή την εγγύηση, ας πούμε, γιατί μειώθηκε το ποσό της εγγύησης κατά 35%. Αυτά και δεν ξεπέρασα τα δύο λεφτά. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Καράς. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση την οποία κάνουμε ως τώρα για το FC2 καθιστά το σημείο εκκίνησης ε, πιο αισθητό σε σχέση και με αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος. Και νομίζω ότι αυτό που είναι καθοριστικό είναι να μην προσεγγίζουμε τα πράγματα λέγοντας ότι εντάξει λειτουργεί μεν, αλλά το μόνο που δεν λειτουργεί είναι το θέμα των δημόσιων ε, λειτουργίων των τραπεζών και το θέμα των ε, κυβερνήσεων. Όχι. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της διάθρωσης ε, των εργών, των συζητήσεων και να μιλήσουμε σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα όταν ούτε οι οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ξέρουν πώς να ενημερωθούν και ποια έργα στη χώρα τους χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΥ, ε, πού το ξέρουν οι τοπικές ε, αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ενημερωθούν τα τοπικά κοινοβούλια, το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα να έχουν οι βουλευτές τη δυνατότητα να ενημερώνουν τον υπόλοιπο κόσμο για τις επιτυχίες του FC. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Το θέμα του ΕΦΣΙ για μένα δεν είναι θέμα μόνο του κατά πόσο οι τράπεζες χρησιμοποιούν την χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ. Το βασικό θέμα είναι αν έχουμε τόσα πολλά έργα από την ιδιωτική οικονομία ώστε να είμαστε στο Champions League των επενδύσεων και έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε πολύ λίγο equity και έχουμε ακόμα πολύ λίγη συμμετοχή από το εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους... στον κύριο Κορυμέλα. Δύο λεπτά παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσίαση αυτή. Με ενδιαφέρον σημείωσα τα ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά αυτά αριθμητικά στοιχεία που μας δώσατε για τις υποδομές. 200 ε, περίπου τέτοια εγχειρήματα, 21 τέτοια, τέτοιες πλατφόρμες επένδυσης και το καθεξής. Αλλά να σας πω ότι αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία. Το θέμα είναι, και αυτό το συζητάμε συνέχεια, τι κάνουμε τα χρήματα αυτά. Εσύ μας λέτε ότι είμαστε επιτυχείς επειδή καταφέρουμε να ξοδεύουμε τόσα εκατομμύρια ευρώ. Ε, εγώ το να σας πω, το πιστεύω ότι αυτό λίγο πολύ όλοι μπορούν να το κάνουν. Δεν νομίζω ότι αυτό μας κάνει ιδιαίτερη στους Ευρωπαϊκή Ένωση, το τα ξοδεύουμε τα χρήματα. Αυτό που θα μας έκανε ξεχωριστούς θα ήταν να πετύχουμε το στόχο του προγράμματος μία συμπληρωματικότητα, η οποία δεν θεωρώ ότι αποδεικνύεται πουθενά σε καμία περίπτωση. Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι πολλοί από τους ομιλητές διαπίστωσαν πόσο επιτυχές είναι το εύση στην ομιλία τους, στην παρέμβασή τους και ουσιαστικά θέτουν το ίδιο ερώτημα όπως εγώ. Μα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις κρίσεις μας και στην αξιολόγησή μας. Να περιμένουμε πρώτα συγκεκριμένα αποτελέσματα, πρωτού κρίνουμε κατά πόσο ήταν επιτυχές ή όχι το ΕΦΣΥ. Το θέμα λοιπόν είναι πού είναι η σκοπιμότητα των έργων, πώς μπορεί να καταμετρηθεί, πώς μπορεί να καταμετρηθεί ο αντίκτυπός τους, πού βρίσκεται η προτιθήμενη αξία στο δημόσιο τομέα, γιατί στο δημόσιο τομέα είναι σαφές ότι ό,τι περνάει από το ΕΦΣΥ αποτελεί ή μία νέα χρέωση ή ουσιαστικά καταπίεση ήδη φυστάμενων έργων. Έχω στρατηγικό πώς προβλήματα με αυτά που σας αναφέρω και θα ήθελα διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να δώσω το λόγο τώρα στον Σάντερ Λόντς. Και θα τον αντικαταστήσει υπάρχει κάποιος. Όχι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Νίλ Στόρβαντς από το Άλντε. Ή μάλλον ε, η κυρία Γκουλάχ θα τον αντικαταστήσει. Θα μπορούσε ίσως να μιλήσει και εξ ονόμας του κυρίου Ραμόν Τρεμόζα. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τρεμόζα. Α, Σιλβί, μίλησε. Λοιπόν, πες ό,τι θέλεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λοιπόν. Εκ μέρους του Νίλς. Σύντομα, η Άντε είναι υπέρ της παράτασης του ΕΦΣΥ και της χρηματοδότησης, αλλά δεν μας αρέσει η πρόταση να περικόψουμε το Connecting Europe Facility. Ε, ε, αν γίνουν και άλλες περικοπές, πολλοί προβουλευτές είπαν ότι δεν θα το εγκρίνουν. Ε, η μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του, ΚΑΠ, του COP21 είναι πολύ θετικό πράγμα καθώς και το παράθυρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να διευκρινίσει ε, τι γίνεται με την ηχθειοκαλλιέργεια, ε, γεωργία και ηχθή και αλία, ότι είναι εντός του ΕΦΣΥ. μιλάμε για τον τίτλο 1α, χρηματοδότηση δηλαδή από την εγγύηση του ΕΦΣΥ. Η συζήτηση εντός της Κομισιόν ε, πώς εξελίσσεται για αυτό το θέμα. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάτι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ευρύτατη προσέγγιση. Ήταν καλή αυτή η πρωτοβουλία, το ΕΦΣΥ, βοήθησε να εξασφαλίσουμε περισσότερες επενδύσεις, αλλά ο λόγος που δημιουργήθηκε ήταν ότι ήταν δύσκολο οι εταιρείε να βρουν τελικά χρηματοδότηση από τις αγορές. Σας κάνω έκκληση να προωθήσετε την Ένωση Κεφάλαια Αγορών και ούτως ώστε να προχωρήσουν όλα αυτά, αυτοί οι φάκελοι να προχωρήσει το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν έχω μια τέτοια ε, συνεκτική προσέγγιση, θα φτιάξουμε ουσιαστικά πακέτα όπου θα βρούμε, όπου θα βρούμε συμφωνία. Αυτά, καλή τύχη και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστούμε Σιλβί. Τώρα, κανονικά θα πρέπει να πάρει το λόγο ο κύριος Ριάντα από το Badge. Νέα Επιτροπή Μπάτζ, προπολογισμού δηλαδή. Δεν τον βλέπω. Ποιο θα τον εκπροσωπήσει από την ΚΟΕ. Έχετε δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα, η θέση μας καταρχάς σε σχέση με αυτό το σχέδιο. Εμείς θεωρούμε πως δεν είναι παρκές ε, για να υπάρξει ανάκαμψη. Θα έπρεπε να υπάρξει ένα πραγματικό σχέδιο δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, ε, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει χρήματα στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ε, στο πλαίσιο του Quantitative Easing, AXA, Total, Lucid, Daimler και ένα σωρό άλλες εταιρείε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και που είναι σημαντικά στην υπηρεσία ενός πραγματικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που θα ήταν πολύ πιο απλό και πιο αποτελεσματικό. Εγώ έχω μια ερώτηση σε σχέση με τα νούμερα που μας παρουσιάσατε. Ε, ότι, λέει η αξιολόγηση ότι η Πορτογαλία είναι μια από τις χώρες που περισσότερο ωφελήθηκε και από το σχέδιο Juncker. Από όσο εμείς γνωρίζουμε, σε αυτή τη φάση συγκεκριμένα υπάρχει μία επένδυση του, του Δήμου της Λισαβόνας, 50, ε, 500 εκατομμύρια ευρώ λέει, αλλά συγκεκριμένα Πρόκειται για ένα δάνειο 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμή. Ήταν έναν 100 ε, δισεκατομμύρια και ο Δήμος έκανε πίσω και ε, ε, τελικά κατέληξε σε ένα δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν συμφωνίε με ένα σύνολο τραπεζικών θεσμών που θα χρηματοδοτήσουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Εμεί όμω δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τι επενδύσει επιτόπου. Ε, και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Έπειτα, υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση του ίδιου του ταμείου. Δηλαδή υπήρχε στην ουσία ένα μενού ε, ε, επενδύσεων και οι επενδυτές θα διάλεγαν από αυτό το μενού. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν πέρα από τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Τράπεζας Επενδύσεων, ποια είναι η, ποιος είναι ο ισολογισμός της εξωτερικής δράσης των ιδιωτών, που, είτε των χωρών είτε των ιδιωτών επενδυτών. Στην πραγματικότητα έχω δύο ακόμα λεπτά να κάνω και άλλη μια παρέμβαση μετά που θέλω να προχωρήσω. Ναι, να προχωρήσω. Μάλιστα, το δεύτερο μου ερώτημα λοιπόν αφορά την, το κατά πόσο όντω υπήρξαν αυτές οι, ε, οι επενδύσεις. Ναι, ναι, εγώ τον αντικαθιστώ, οπότε είναι εντάξει το Φάβιο Ντεμάση. Ε, λοιπόν, Δεύτερη μου ερώτηση αφορά την υλοποίηση των επενδύσεων. Τρίτη μου ερώτηση έχει σχέση με την γεωγραφική κατανομή. Εμείς εδώ είμαστε εμπερδεμένοι και προσπαθούμε να φτιάχνουμε διαφόρους μηχανισμούς που μέσα από την αξιολόγηση των επενδύσεων βλέπουν αν λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική κατανομή και αν τελικά οι περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση, εδώ δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι μάλλον περισσότερο διαπίστωση ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πρέπει να είναι πολύ ε, πιο απλά τα πράγματα να διατηρηθεί ένα κομμάτι αυτού του σχεδίου με κριτήρια γεωγραφικής κατανομής ε, αντί αυτή τη στιγμή να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να επιβάλλουμε κριτήρια κατόπιν εορτή στο Συμβούλιο Αξιολόγησης των Επενδύσεων. Και η τελευταία ερώτηση αφορά ένα άρθρο το οποίο διαπίστωνε, εξέταζε μάλλον τον κανονισμό. Ένα άρθρο μάλλον του κανονισμού που, που έλεγε ότι θα δοθεί παράτωση μετά από μία ανεξάρτητη εξολόγηση. Δηλαδή, να δούμε ε, από, αν έγιναν οι επενδύσεις, αν έγιναν με διαφάνεια, αν έγιναν ε, σωστά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται τον κανονισμό που έχουμε εγκρίνει εμείς εδώ και που υποχρέωνε στην υλοποίηση μιας ανεξάρτητης ε, αξιολόγησης του Ταμείου και πώς αυτό λειτουργήσε. Για ποιους ακριβείς λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δοθεί παράταση χωρίς να γίνει αυτή η προβλεπόμενη αξιολόγηση. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Θα δώσω τώρα την Προεδρία. 45 λεπτά πέρασαν στον Συμπρόεδρο της ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εξ των Πρασίνων, Σολέ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΕΦΣΙ είναι εν γέννη καλό πρόγραμμα, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ωστόσο, θεωρούμε πως είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση του ΕΦΣΙ, ακριβώς επειδή ε, δεν έχει λειτουργήσει αρκετό καιρό ώστε να μας μπορέσουμε να κάνουμε αξιολόγηση ποσοτική και ποιοτική. Δεύτερον, θεωρούμε ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την επιλεξιμότητα, αλλά και ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για την διαφάνεια. Ιδιαίτερα όσον αφορά την προσθετικότητα των project και την συμβολή στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όσον αφορά τι επενδύσει προσθετικότητα, αυτέ θα πρέπει να είναι πάντοτε σύμμορφε προ τι στρατηγικέ ανάγκε τη ευρωπαϊκή οικονομία. Μία εξ αυτών είναι, για παράδειγμα, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Επίσης θα πρέπει το ΕΦΣΙ να γίνει πιο προσιτό στις μικρομεσαίες γιατί όπως γνωρίζετε αυτές είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και το κατόφλι των 25 ε, εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να χαμηλώσει και θα πρέπει να είναι ευκολότερο να δημιουργηθούν πλατφόρμες επενδυτικές. Και ως προς αυτό ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να προωθήσει την προσέγγιση των επενδυτικών αυτών πλατφορμών και για άλλα project που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκάουτ, από τους πράσινους, από την ΕΚΟΝ όμως. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Χρειάστηκε να πάω και στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Προς πίσω πάω. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος το εξής. Έχω την αίσθηση ότι όλοι λένε «Οκ, okay, μια χαρά, καλό είναι το ΕΦΣΙ, πρέπει να το βελτιώσουμε και να συνεχίσουμε». Αλλά ξέρω ότι το ελεγκτικό συνέδριο ήταν πολύ πιο επικριτικό και ουσιαστικά λέει ότι δεν υπάρχει λόγος για, παράτασης, για παράταση του Εύση, λόγω του πώς ε, τα έχει πάει μέχρι τώρα. Αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη και να εξασφαλίσουμε ότι οι βελτιώσεις που κάνουμε δικαιολογούν την παράταση του ΕΦΣΥ, γιατί συμφωνούμε απόλυτα ότι ένα πρόγραμμα επενδύσεων σίγουρα χρειάζεται, αλλά το να το κάνουμε με δημόσια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός είναι ο τρόπος ε, και να εξασφαλίσουμε ότι η προστατικότητα είναι πραγματικά επιπρόσθετη και ότι ε, συνάδει απόλυτα με τους στρατηγικούς μας στόχους. Αυτό σημαίνει προστατικότητα και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που κάνει το ΕΦΣΥ πάνε εκεί όπου δεν θα γινόταν χωρίς το ΕΦΣΥ, δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς το ΕΦΣΥ. Τώρα έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει αυτά που κάνει πάντα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν πρέπει να συμβαίνει όμως αυτό. Δεν παίρνει δημόσιο χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τα ίδια με παλιά. Αυτό είναι σημαντικό. Μερικέ από τις αλλαγέ και τις βελτιώσεις που, που εξασφαλίζει η Κομισιόν ε, μερικές φορές μας δημιουργούν ερωτηματικά, α πούμε για το κλίμα. Λέμε project με συνιστώσει που συνεισφέρουν στην κλιματική δράση. Τι είναι αυτό. Δεν είναι σαφές ότι υπάρχει προστατικότητα εδώ. Εμείς θέλουμε project αποκλειστικά για την κλιματική ελέγχη που δεν υπάρχουν ακόμα. Δεν θα πω και πολλά ακόμα. Αυτό που θέλω όμως είναι να υπάρξουν βελτιώσεις του ΕΦΣΥ και να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πραγματικά ε, προσθετικότητα και όχι, δεν παρατείνουμε απλώς το ΕΦΣΥ έτσι, χωρίς κανένα στόχο. Ο Μάρκο Βάλλη από την ΕΚΟΝ, η FDD. Ευχαριστώ. Καταρχάς, κάτι θεμελιακό. Αν πολιτικός πώς θέλουμε να ξαναδρομολογήσουμε τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε να τονώσουμε την ζήτηση. Ένα σχέδιο όπως αυτό του Juncker ή όπως το ΕΦΣΙ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει αυτό που χρειαζόμαστε αυτό που χρειάζεται η οικονομία μας. Δηλαδή, λείπει το δημόσιο χρήμα. Σημαντικά δημόσια κονδύλια. Δεν αρκεί μια τόσο μικρή εγγύηση για να δρομολογηθεί εκ νέου η οικονομία. Και με ανησυχούν τα δεδομένα που δίδονται, γιατί είναι μια στιγμή όπου τα δεδομένα είναι διωγγωμένα και από το quantitative easing που κράτησε χαμηλά την αξία του ευρώ και από την τιμή του πετρελαίου που πριν από λίγο καιρό ήταν πολύ χαμηλή η τιμή του. Είναι μια ανάπτυξη βέβαια, αλλά που δεν θα είναι ε, μακροπρόθεσμη. Και πολύ γρήγορα θα, επανα... θα ξαναεμφανιστούν τα παλιά και γνωστά προβλήματα της ε, Ευρωζώνης. Εάν δεν τονώσουμε περισσότερο τη ζήτηση, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το πρόβλημα τη προσθετικότητα που το ανέφεραν πάρα πολύ, θέλουμε να μάθουμε το εξή. πώ στο εσωτερικό τη Κομισιόν, αν βλέπετε, που βλέπετε τα διάφορα project και εντό του υπάρχουν διάφορε πληροφορίε, αλλά λείπει ε, μία ανεξάρτητη αξιολόγηση πραγματικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δίνω, δώσουμε εξήγηση στου πολίτε, γιατί, παραδείγματο χάρη, ε, προωθούμε ας πούμε μία πλατφόρμα πετρελαίου ή ένα αυτοκινητόδρομο ας πούμε ε, που θα έπρεπε να έχουν ε, σημαντική, που έχουν μάλλον σημαντική περιβαλλοντική αξία. Αλλά δεν υπάρχει ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση και μόνο η Κομισιόν μας δίνει τις πληροφορίες ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν αρκεί αυτό γιατί οι πολίτες δεν πείθονται ας πούμε, ότι αυτά τα project ας πούμε, κάνουν τη διαφορά ε, ας πούμε, ένα δηληστήριο ή οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανεξάρτητη διαλόγηση για να ξέρουμε για ποιους λόγους ε, προωθούνται κάποια project και κάποια όχι. Ε, Μάρκο Ζάνη, από το ENF, Badge. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω να πω και πολλά για αυτή την πρόταση της Κομισιόν που τη βλέπω ανεξήγητη. Δεν καταλαβαίνω. Και ο συνάδελφος από τους πράσινους προηγουμένως μίλησε για το για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Διαβάζοντάς τη βλέπετε ότι δεν είναι σαφές αν πετύχαμε κάποιον από τους στόχους. Μετά από 1,5 χρόνο λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε ότι χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις ενός προγράμματος που θεωρείται τόσο σημαντικό, έκτακτο, όχι συνήθες κτλ. Η Κομισιόν χωρί αξιολόγηση προτείνει την παράτασή του. Ή τέλο πάντων ε, υπό λιγάκι διαφορετική μορφή. Λείπει η διαφάνεια, λείπουν τα στοιχεία, τουλάχιστον για μένα, για να αξιολογήσω τι επιπτώσει αυτής της πρώτης ε, φάσης. Η πρώτη έκθεση που μα ε, έφτασε είχε στοιχεία αλλά όχι λεπτομερείς. Για, για το 90% των περιπτώσεων δεν καταλαβαίνουμε με ξεκάθαρο τρόπο Ποια είναι η προσθετικότητα, αυτή η προσθετικότητα πούμε, που θεωρείται βάση, ο επιλώνας ε, αυτού του εύση, δεν προκύπτει. Δεν υπάρχουν πληροφορίες λεπτομερείς για την επίπτωση που έχουν αυτά τα project ή είχαν στην οικονομία των κρατών μελών ή των περιφερειών όπου υλοποιούνται. Και δεν υπάρχει ε, ασφάλεια για το πολλαπλασιαστικό τους χαρακτήρα. Το είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Η Κομισιόν μίλησε για να πολλαπλασιαστεί και έφτασε σε αυτό το νούμερο των 170 δισεκατομμυρίων και που μας είπατε. Αλλά ε, το, το ελεκτικό συνέδριο είπε ότι δεν υπάρχει σιγουριά. Ότι πρέπει να ξαναδείτε το πώς, τη μεθοδολογία με την οποία ε, χρησιμοποιείται αυτό το πολλαπλασιαστή. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ας πούμε, όπου έγιναν λάθη με τα νούμερα. Όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με τα νούμερα. Αν χρειάζεται, ας βρούμε περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουμε τι πετυχαίνει σήμερα, τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα το ΕΦΣΙ. Και ας βρούμε το χρόνο, τόσο ώστε αυτή η πρωτοβουλία και η παράταση του ΕΦΣΙ να μην θεωρηθεί ως προπαγάνδα προπαγανδιστικό κίνημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που βρίσκεται εκεί στην, στην κοσμάρα της. Γιατί δεν βλέπω ε, αποτελέσματα ακόμα. Α, συγκεκριμένα. Και όσο περισσότερα μου λέει η Κομισιόν, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι στην πραγματικότητα είναι ένα προπαγανδιστικό, μια προπαγανδιστική κίνηση. Αλλά θα σας δώσουμε πιο πολύ χρόνο, πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι δικαιούστε. Και τώρα λοιπόν θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Τέσσερα μέλη έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μάλετιτς από την Επιτροπή ΕΚΟΝ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί το ΕΦΣΥ. δεν είναι το θέμα μόνο η χρηματοδότηση, αλλά και οι υπόλοιποι πυλώνες που συνδέονται με την καλή εφαρμογή του ΕΦΣΥ ως ταμείο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την ενιαία αγορά, τις μεταρρυθμίσεις, τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να υπάρχει μια δρομολόγηση των έργων με καλό σχεδιασμό και θετικό αντίκτυπο τελικά και για το ΑΕΠ και τι θέσει απασχόληση. Μιλήσατε για τη Ρουμανία, ότι υπάρχει έλλειψη έργων με σωστή προετοιμασία και με σωστή κατάρτιση και διάρθρωση των έργων. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν συμμετέχουν. Όχι σε ικανοποιητικό επίπεδο τουλάχιστον στο ΕΦΣΥ. Και ίσως η διαφάνεια αυτή να πρέπει να επικεντρωθεί στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ κρατών μελών. Καλών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Για να βοηθηθούν οι χώρες που δεν έχουν ακόμα συμμετάσχει στο σωστό επίπεδο. Μιλάμε για το blending, την ε, μεικτή χρήση τέτοιων χρηματοδοτικών κονδυλίων. Αυτό δεν λειτουργεί ακόμα σε σωστό επίπεδο, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε. Άλλοι είναι οι κανόνε για το ορίζοντα 2020, άλλοι το ΕΕΦΣΙ, άλλο για το τα ταμεία. Και ιδιαίτερα θα μιλάμε για κρατικέ επιδοτήσει και κάποια άλλα σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, και σα παρακαλώ. Το η συναδελφοί, ένα λεπτό διαρκεί. Σα παρακαλώ, μην ε, μακρηγορείτε. Ο κ. Μαρινέσκου από την Επιτροπή Ελέγχων Προεπιλογισμών από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για το παράδειγμα που δώσατε για τη Ρουμανία. Αληθεύει όντω το γεγονός ότι μόνο ένα έργο έχει υπογραφεί στην Ρουμανία και έχουμε και κάποια άλλα τα οποία έχουν λάβει έγκριση ή προέγκριση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε γιατί δεν υπάρχει καμία τράπεζα προώθησης εκεί. Γιατί οι τράπεζες από τη Ρουμανία, οι τράπεζες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, που κάνουν συναλλαγές στην Ρουμανία, ε, ασχολούνται με το έψη στις χώρες τους, αλλά όχι στη Ρουμανία. Και γιατί δεν υπάρχει κόμμος λοιπόν στη Ρουμανία, γιατί αυτό θα χρειαζόταν και σε ό,τι αφορά την διαφάνεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Να δούμε γιατί εγκρίθηκε ή δεν εγκρίθηκε μια αίτηση, τα κριτήρια για την συμπληρωματικότητα να τα δούμε και για τις μικρομεσαίες. Νομίζω ότι σημασία έχει να δούμε επίσης πόσα χρήματα φτιάχνουν, φτάνουν τελικά στους δικαιούχους και πόσα χρήματα φτάνουν τελικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πιστεύω ότι ίσως να μεταφραστεί και επιτέλους αυτή η ιστοσελίδα του ΕΦΣΙ και στα ρουμάνικα. Δεν υπάρχει ρουμάνικη μετάφραση. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε μια παρουσίαση σε 100 άτομα για το ΕΦΣΙ σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε πιο πολύ. The third one Η κυρία Χόλμαϊερ Κύριε Αντιπρόεδρε, καταρχά να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σα. Αυτό που θα με ενδιαφέρει εμένα θα ήταν το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει λίγο πιο πολλέ πιστώσει και λιγότερε επιδοτήσει. Και συμφωνώ όταν πρόκειται για έργα τα οποία είναι κοντά στην αγορά. Αλλά όταν πρόκειται για έργα τα οποία είναι πιο πολύ του ορίζοντα 2020 και έχουν να κάνουν με την έρευνα, την διαθυμηματική έρευνα. Πιστεύω ότι αυτό δεν υποκαθιστάται από, την, από κάτι άλλο. Έχουμε επαφές και με πανεπιστημιακά ιδρύματα και με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και μας λένε ότι όταν δεν υπάρχει επιδότηση δεν θα προωθηθούν και κάποια συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν να προσέξουμε να δίνουμε πιο, πολλά, πιο πολλές ε, ε, επιδοτήσεις σε τέτοια έρευνα η οποία δεν είναι τόσο κοντά στην αγορά. Αυτό να το αφήσουμε για το ΕΦΣΥ. Αυτή την απόπειρα να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν με καλωρίσετε κιόλα, λέει ο Πρόεδρος. Από την οίκον Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Φρουντζούλικα. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως η παρέμβαση του Αντιπρόεδρου Κατάινεν, ε, ξέρετε, είναι ένα παράδειγμα, έδωσε τη Ρουμανία και γι' αυτό δεν μπορούσα να πάρω το λόγο το ΕΦΣΥ. Έχει πραγματικά αποδώσει πέραν κάθε προσδοκία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περισσότερες χώρες. Δεν καταλαβαίνουμε όμως γιατί δεν το πετύχαμε αυτό στη Ρουμανία, γιατί εγώ ε, συμμετείχα σε διάφορες οργανώσεις. Υπάρχουν χιλιάδες, χιλιάδες, πολλές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση για πιστώσεις, για εγγύησεις. Ε, πάνε στις τράπεζες και οι τράπεζες λένε πως δεν ξέρουν καν το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Οι τράπεζε λένε πω οι δικέ μα μικρομεσαίε δεν ενδιαφέρονται. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχουμε εξαιρετική υγεία και παρά, παρόλα αυτά εισάγουμε πάνω από 70% των γεωργικών προϊόντων λόγω έλλειψη χρηματοδότηση για μικρομεσαίε ε, επιχειρήσεις που δουλεύουν τη γεωργία. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν, γιατί κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου να σα πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο φόβο που επικρατεί στη χώρα μου και το έχω δει και σε άλλε χώρε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ότι δηλαδή μετά από όλε αυτέ τι ε, ανακοινώσει με, για ε, την ευρωπη δυο δύο-τριών ταχυτήτων ο κόσμος ανησυχεί, φοβάται ότι θα πέσουμε σε κάποια φαιά περιοχή αβεβαιότητας και φόβου. Και κάτι πρέπει να γίνει ώστε να διατηρηθεί η ενότητα της Ευρώπης για το μέλλον, γιατί διαφορετικά αυτό θα είναι ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη που θα γεννηθεί πάλι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να κρατάτε το χρόνο που σας έχω δώσει. Μπέρες κυρία Μπερές, παρακαλώ, ένα λεπτό που είστε συντονίστε της ΕΚΟΝ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριε την Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση που ήδη έχει τεθεί πάνω κάτω και είναι το θέμα του μακροοικονομικού αντίκτυπου του ΕΦΣΙ, διότι στη φάση αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να επαληθεύσουμε αν όλα τα συστατικά που θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να βάλουμε μάλλον στο σχέδιο και στην αρχή, υπάρχουν ακόμα. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι, και δεν επανέρχομαι στο θέμα της προσθετικότητας γιατί είναι πολύ συζητημένο, τι θα πρέπει να βελτιώσουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτό ώστε να είναι πιο προσιτό και πιο γνωστό. Θα θυμάστε με, με τον Κριστιαν Ελέρε αγωνιστήκαμε ώστε οι ε, πολιτιστικές και δημιουργικές ε, επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και αυτές από τα ΕΦΣΙΑ. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος που να πάει να τους βρει, να τους πιάσει από το χέρι και να τους δείξει πώς θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση, δεν θα γίνει ποτέ. Οι δομές προώθησης του ΕΦΣΙ που έχουν στηθεί είναι σωστές, είναι και πώς μπορούν να βελτιωθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάρη από το Έκον. Η κυρία Καϊλή με συγχωρείτε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα για το FC2. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το θέμα της διαφάνειας που χρειάζεται ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα project που έχουν ιεραρχηθεί είναι αυτά που δεν μπορούσαν να πάρουν χρηματοδότηση από άλλους πόρους, δηλαδή υπογραμμίζω την ανάγκη προσθετικότητας. Επίσης να έχουμε πιο πολλά διασυνοριακά project. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό γιατί ένας από τους στόχους μας ήταν να μειώσουμε τις ανισότητες ανάμεσα στις χώρες και αυτό ε, θεωρήθηκε καλό εργαλείο για την επιτευχή αυτού του στόχου. Κάτι ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε χώρα δεν θα ε, ωφεληθεί πάνω από το 10% του ΕΦΣΥ στο σύνολο, ώστε να μην ε, επικεντρωθεί το, η χρηματοδότηση μόνο σε μια χώρα. Μια χώρα 10% στο σύνολο, 50 δις νομίζω, είναι, ακριβά, είναι αρκετά χρήματα που, ώστε να έχουν αντίκτυπο γιατί πρέπει να διορθώσουμε και όχι να αυξήσουμε τη διαφοροποίηση στον επενδυτικό χάρτη της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει ίσως να διορθώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την επιτυχία. Γιατί αν μια χώρα έχει ήδη λάβει λιγότερο από ένα δις από τα 170 θεωρείται επιτυχία. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Κατάινεν Τελευταία μας ομιλητή στο ΚΑΤΣΔΙ είναι η κυρία Μποναφέ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα εγώ πιστεύω πως αν θέλουμε να δώσουμε μια αντικειμενική κρίση για το ΕΦΣΙ πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα γεγονός, δηλαδή το μεγάλο χάσμα επενδύσεων στην Ευρώπη και να δούμε πώς αυτό το μέσο θα, θα χρησιμοποιηθεί σωστά. Είναι καλό το μέσο με κάποια όρια, αλλά καλό, θετικό. Όπως είπαν κάποιοι που προηγήθηκαν, είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη δυσκολία για τις επενδύσεις είναι το να ε, κινητοποιηθούν οι πόροι στην αγορά. Και εδώ θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει πολύ σοβαρές και αποτελεσματικές δράσεις στις, ε, ε στην Ένωση Κεφαλαγορών και την Τραπεζική Ένωση. Επίσης, ε, το ερώτημα που θέλω να θέσω στην Κομισιόν είναι Έχουμε στοιχεία για τις θέσεις αποσχόλησης επιπλέον που δημιουργήθηκαν σε σύγκριση με τα χρήματα που έχουν επενδυθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα έχουμε τους τελευταίους ε, που έχουν ζητήσει το λόγο στο Catch Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Φυσικά αύριο και πιο μετά, μέσα στην εβδομάδα η Τερίζα Μέη η Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου θα επικαλεστεί το άρθρο 50 και τμήμα του ΕΦΣΥ, θα, μάλλον τμήμα των αντιπραγματεύσεων θα είναι και το ΕΦΣΥ, αυτό περιλαμβάνει 5 δις. Πείτε μας, τι ποσοστό των 5 δις αυτό έχουν εκχωρηθεί για το Ηνωμένο Βασίλειο από τα 60 δις εγγύησης. Τι ποσοστό αναλογεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέλος όταν κοιτάμε τα project, τα έργα. Έργα όπως για παράδειγμα επενδύσεις 200 ε, εκατομμυρίων θα υπάρχει μία λίστα για τους διαπραγματευτές ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο που θα εντοπίζουν όλους τομείς ε, τους οποίους έχουν στην ιδιοκτησία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και να δούμε στις διαπραγματεύσεις τα νεκτήματα και τα πλανεκτήματα ποιος θα πάρει Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γούλφ ήταν αυτός από τους μη εγγεγραμμένους. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κατάινεν για να συνοψίσει και να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ καλές ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία για το τι είναι το μερίδιο της του Ηνωμένου Βασιλείου για τη χρήση του κεφαλαίου. Αν με ρωτάτε, να κάνω μια εκτίμηση, θεωρώ ότι έχει ωφεληθεί πολύ παραπάνω τον νεμένο Βασίλειο από ό,τι έχει δώσει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Θεωρώ ότι τα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσά, είναι πολύ περισσότερα από την πλευρά των συν παρά των πλην αυτά, για τα θέματα της συμπληρωματικότητα. Όπως είπαν όλοι, αυτή είναι η καρδιά, ο πυρήνα όλου του εγχείρηματο. για την αναθεώρηση εν πάση περιπτώσει, για το fc 2.0. Η ιδέα είναι όλα τα έργα τα οποία εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξηγείται γιατί έχουν επιλεχθεί. Και γιατί χρηματοδοτείται το κάθε έργο από το ΕΦΣΥ προκειμένου όλοι να κατανοήσουν κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχουμε θέσει και στον πίνακα και από πού προέρχεται η συμπληρωματικότητα και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα. σημαντικό και για σας αλλά σημαντικό και για τον υπόλοιπο κόσμο να ξέρουμε τι είδου έργα τελικά παίρνουν χρηματοδότηση και μετά να δούμε αν χρειάζεται ενδεχομένω να αλλάξουμε τον κανονισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το θέμα της διαφάνειας είναι κέρια σημασία. Τώρα, για την έλλειψη ενημέρωση. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό, γιατί είπατε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Ο κύριος Μαρινέσκου έδωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το τι θα πρέπει να συμβεί σε βασικό θεμελιώδες επίπεδο. Όπως σας είπα, πολλοί βουλευτές έχουν οργανώσει εκδηλώσεις ε, για να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες, με τις τοπικές αρχές. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κρατημέλη έχουν επίσης οργανώσει πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, η Ισπανία, η Ιταλία και η Σλοβακία κυρίως. Έχουν δηλαδή προσπαθήσει να εξηγήσουν και σε απομακρυσμένε περιοχές, στι επιχειρήσεις και στου ηθήνοντε, το πώ λειτουργεί το ΕΦΣΥ. Για το μακροοικονομικό αντίκτυπο και για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργήσε το ΕΦΣΥ. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή αριθμητικά στοιχεία, αλλά η ΕΤΕΠ μας υποσχέθηκε κάποια πρώτα αποτελέσματα για το ΕΦΣΥ και τις θέσει εργασία. Αλλά είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι άμα υπάρχουν ήδη 400.000 επιχειρήσεις που ωφελούνται, ε, τι δουλειέ συνεπάγεται αυτό, πόσε θέσει απασχόληση, δεν ξέρω. Μία αναεπιχείρηση, δύο αναεπιχείρηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, α μην τριαμβολογούμε ακόμα πριν λάβουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η ΕΤΕΠ. Η ΕΤΕΠ δεν συνεχίζει business as usual. Χρηματοδοτούν πιο πολλά πιο πολλά μετοχικά προγράμματα, πιο πολλά προγράμματα equity και έχουν πιο στενέ επαφέ με τι εθνικέ τράπεζε από ό,τι είχαν ε, παλιότερα από πλευρά τη ΕΤΕΠ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή παύλα γεωγραφική κατανομή. Μία από τις προτάσεις στην αναθεώρηση του ΕΦΣΥ είναι να επιταχυνθεί η τεχνική αρρωγή επιτόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΤΕΠ θα δίνει πιο πολλούς ανθρώπινους πόρους προς την κατεύθυνση αυτή. Η ΕΤΕΠ επίσης έχει συμφωνήσει για την τεχνική αρρωγή επιτόπου. Πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ενημέρωση. Και όπω είπατε, αυτό μερικέ φορές μπορεί να είναι περίπλοκο, για γραφειοκρατικούς δηλαδή λόγου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνει τέτοια ανάμειξη των χρηματοδοτικών κονδυλίων, αυτό το blending για τις πλατφόρμες τώρα. Αυτό σίγουρα αποτελεί μία προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε πιο πολλές πλατφόρμες για τους λόγους που αναφέρετε όλοι σας. Ένα θετικό παράδειγμα να σας δείξω για πλατφόρμες. Ο συναδελφός Σεύκοβιτς και ο κύριος Κανιέτε δημιουργούν πλατφόρμες ενεργειακής αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας ε, τα δραστηριακά ταμεία από κοινού με το ΕΦΣΥ. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Και μερικοί εξημών θα γνωρίζετε την πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η ιδέα για τι μικρομεσαίε λοιπόν επιχειρήσει, θα μεταφερθεί για την ενεργειακή αποδοτικότητα και έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται διαφορετικά ταμεία μαζί με το ΕΦΣΥ για ενεργειακά έργα. Για τη Ρουμανία τώρα. Όπω σα είπα, η κατάσταση θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αλλά και σίγουρα θα βελτιωθεί στο μέλλον. Γι' αυτό είμαι βέβαιο. Σε κάποιε περιστάσει πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ενδιαφέρουσε προκλήσει στα κράτη-μέλη. Δύο παραδείγματα επιτρέψτε μου. Για την Ελλάδα και για την Ρουμανία. Υπάρχει ένα έργο στην ε, Ρουμανία για την ε, άρδευση με χρήση του Δούναβη. Ήταν ένα από τα μεγάλα, μεγάλα τέτοια έργα στη Ρουμανία όπου ενδεχομένω να γινόταν χρήση του Εύση. Αλλά είχαμε την εντύπωση ότι επειδή το ΕΦΣΙ δεν δίνει επιδοτήσεις, δεν ενδιαφέρθηκε η κυβέρνηση της Ρουμανίας για το ΕΦΣΙ. Τα νομικά συστήματα στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά άκαμπτα. Δεν επιτρέπουν να προχωρήσουν γρήγορα τέτοια πρόγραμματα. Ένα άλλο παράδειγμα από την Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε τις ελληνικές αρχές προκειμένου να δημιουργήσουν ε, πλατφόρμες ε, δημοσίου και ιδιωτικού σύμπραξης και δημοσίου τομέα, όπου οι αρχές θα μπορούσαν να συνδυάσουν τα αγροτικά ταμεία με το ΕΦΣΥ και με κάποια ιδιωτικά κεφάλαια. Και αυτό θα αποτελούσε εξαιρετικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου είχαν μεγάλα προβλήματα σε χρηματοδότηση από πλευρά των τραπεζών. Παρά το γεγονός όμως ότι προσπαθήσαμε σκληρά να βοηθήσουμε, ώστε δεν έχουμε πετύχει. Ε, εντάξει, πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειε, αλλά να πω ότι σε κάποιες περιστάσεις, περιπτώσεις είναι πολιτικός πως δύσκολο να έχουμε καλές λύσεις. Κι άλλο ένα θέμα. για την ενημέρωση των Ευρωβουλευτών για τα έργα. Να επιστήσουμε την προσοχή σας και θέλουμε να σας ευαισθητοποιήσουμε σε ό,τι αφορά τέτοια καλά έργα και επίσης να σας ενημερώνουμε για έργα στην εκλογική σας περιφέρεια για να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις αυτές γιατί είναι σημαντικό και οι επενδυτές αλλά και το κοινό να βλέπουν αναγνωρίσιμα πρόσωπα, όπως είναι οι ευρωβουλευτές σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στέλνει αυτό ένα μήνυμα ότι συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα αυτό και αυτό με τη σειρά του προσευχή μελλοντικού επενδυτές και για άλλα έργα. Τελευταίο σημείο τώρα. Για το Connective Europe Facility έχουμε 17,5 εκατομμυρία και 500 εκατομμύρια για το ΣΕΦ. 1,1 δις έχουμε σε συνδυασμό ΣΕΦ και ΕΦΣΙ. Τα εργαλεία του ΣΥΕΦ είναι πολύ πιο περιπλοκά από ότι αυτά του ΕΦΣΙ. Γι' αυτό θέλαμε να αυξήσουμε τις επιδοτήσεις και να χρησιμοποιήσουμε το Connecting Europe Facility και σε συνδυασμό με το ΕΦΣΙ, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ πιο πολύ τις επενδυτικές υποδομές με βουλευτέ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων και αν έχετε σε καμία, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε ανάγκη διευκρίνηση, στείλτε μου ένα email και προς την ΕΤΕΠ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Μην διστάσετε. Είμαστε εδώ για να σας βοηθάμε. Ιδιαίτερα αν έχετε καλές ιδέες ή αν θέλετε να ενημερώσετε. Ελάτε να μας επισκεφτείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτροπέ Σα ευχαριστώ πολύ και για την άνοιξη αυτή πρόσκληση για ενημέρωση και για την ε, προσπάθεια που καταβάλλατε. Θέλουν το λόγο οι συγητέ για να συνεψηφίσουν ο κύριος Φερνάνδες. Πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι σήμερα εδώ μαζί μας Κάτι που με εντυπωσιάζει είναι το εξή. Ε, αυτό το κονδύλι θέλει να συνδυάσει τις δημόσιες ε, με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η εγγύηση έχει χρησιμοποιηθεί εκεί όπου έχει χρησιμοποιηθεί και έχει φέρει κέρδη, έχει, έχει οδηγήσει σε επενδύσεις και σε απασχόληση. Πολλά project δεν, που δεν θα είχαν αλλιώ υλοποιηθεί, υλοποιούνται. Πώς μπορεί κανείς να είναι κατά ενό τέτοιου ε, ταμείου που δημιουργεί θέσεις απασχόληση, που βοηθάει στην ανάπτυξη και που ε, είναι προφανές, ε, μπορεί να, είναι, να έχουν γίνει και λάθη, αλλά πώς μπορεί κανείς να μην, να, να μην επιθυμεί την ύπαρξή του. Οδηγεί στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορεί να υπάρχει κάποιος που να είναι κατά της ύπαρξης ενός τέτοιου κονδυλίου. Uma preocupação, κύριε vice-presidente da Comissão. Tem uma preocupação μια ε, ανησυχία έχω κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής σε σχέση με τη χρηματοδότηση των εγγύσεων. Το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει με την Κομισιόν ότι δεν θα είχαμε πια ούτε ένα ευρώ τζακιστό από τον ε, χρηματοπιστωτικό μηχανισμό του ΣΕΦ. Και η πρόταση, στην πρόταση της Κομισιόν ε, αφαιρούνται 500 δις από το παράθυρο των χρηματοδοτικών μέσων. Δηλαδή μειώνεται ακόμα μια φορά το ποσό του ΣΕΦ κατά 500 δις. Εμείς ε, νομίζαμε πως το Συμβούλιο κρατάει τον λόγο του. Είχαμε ε, καταλάβει ότι οι συμφωνίες γίνονται για να τηρούνται. Και αν στον κανονισμό αυτό είχαμε πει ότι δεν θα έρθουμε να ξαναγγίξουμε εκείνα τα χρήματα που συναποτελούν την εγγύηση, τότε αυτά τα 500 δις που βγαίνουν από το παράθυρο χρηματοδοτικά μέσα του, της, της διευκόλυνσης διευρύνοντας την Ευρώπη δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Δεν μπορούμε όντω να αφαιρέσουμε 500 δις από αυτό, από το διευρύνοντα την Ευρώπη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεύτερο τώρα εισηγητή, ο κύριο Μπούλμαν. Σα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Ε, κύριε Κατάινεν, μία έκκληση θα ήθελα να σας απευθύνω. Γιατί και οι δύο πλευρές θέλουμε την επιτυχία του ΕΦΣΥ και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Ελπίζω και το Συμβούλιο το ίδιο να επιθυμεί. Το Συμβούλιο δεν μας έχει ξεχυλήσει και με ενθουσιασμό και δεσμεύση το λέω προσεκτικό. Όταν γεννήθηκε το ΕΦΣΥ, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να μην συμμετέχουν, να μην έχουν μερίδιο μέσω των επενδυτικών του τραπεζών, αλλά όχι με ίδιους ε, πόρους. Αλλά ένα πράγμα δεν θα δεχτούμε και καλό θα ήταν να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξηγήσουμε στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αποδεχτεί τα κράτη-μέλη να Αρχίζουν να ασχολούνται στην, με την πολιτική της ΕΤΕΠ. Τους ανήκει η ΕΤΕΠ και παράλληλα να επιμένουν ότι έλαβαν μία απόφαση για το FC2, για την οποία θα πρέπει να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να κάνει μια πολιτική συζήτηση το Κοινοβούλιο για το πώς ένα εξαιρετικό εργαλείο θα μπορέσει τελικά να δημιουργηθεί. Εξαιρετικό θέλουμε να είναι το εργαλείο αυτό. Και όπως είπε ο συνάδελφος Φερνάντες, ε, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό μπορεί να ε, ενοχλεί κάποιους, αλλά αυτό θα λειτουργήσει μόνο, θα προσπαθήσουμε, αλλά θα λειτουργήσει μόνο αν το Συμβούλιο συμφωνήσει να γίνει μια συζήτηση που θα αυξήσει την ποιότητα του ΕΦΣΥ. Αν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπούλμαν, λέει και ο Πρόεδρο. Έχουμε ολοκληρώσει. Θα ήθελα να σα πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Σε τρει μέρε, στι 16 του Μαρτίου, θα έχουμε σε όλε τι γλώσσε το σχέδιο έκθεση. Στι 20 Μαρτίου, παρουσίαση του σχεδίου έκθεση. 23 Μαρτίου στις 4 ε, το απόγευμα η προθεσμία για τις τροπολογίες. 3 ε, Απριλίου στην Ολομέλεια ε, του Στρασβούργου θα κοιτάξουμε τις τροπολογίες και τις εφαρμοστικές έκθεσης και μετά η ψηφοφορία. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος όλους σας, να ευχαριστήσω και τον κύριο Κατάνη που ήρθε να περάσουμε μαζί το βράδυ μας να περάσετε καλά για το υπόλοιπο βράδυ και θα τα ξαναπούμε σε μια συνεδρίαση της Econ ή της Budget. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.